Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματική η τιμή η παρουσία μου εδώ σήμερα ως υποψήφιος επίτροπος στην ανθρωπιστική βοήθεια και την διαχείριση των κρίσεων. Είναι μεγάλη τιμή που προτάθηκα για αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι στην καρδιά των πανανθρωπίνων αξιών. Έχω πλήρη συνέστηση της τεράστιας ευθύνης. Είμαι ενώπιόν σας ως συνάδελφος, ως πολιτικός που απευθύνεται σε πολιτικούς. Δουλειά μας είναι να λαμβάνουμε αποφάσεις. Συχνά δύσκολες, πολύ δύσκολες αποφάσεις. Ένας πολιτικός είναι σε συνεχή πάλι με την ιστορία. Και είμαστε υπόλογοι προς τις επόμενες γενναίες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όραμα, πολιτικό θάρρος και αξιοπρέπεια. Ευθύνη μου είναι να παράσχω ε, την ε, ηγεσία που θα επιτρέψει το όραμα αυτό να γίνει αποτελέσματα επιτόπου. Οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνονται καθημερινά. Συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή, καταστροφές θεμάτων υγείας, απόλυτη φτώχεια και πείνα είναι τα κύρια αίτια της αύξησης αυτών των αναγκών. Το, τα τρομερά γεγονότα καταδεικνύουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι το τέλος του 2013, 51 εκατομμύρια άτομα ήταν εσωτερικοί εκτοπιστέντες λόγω συγκρούσεων και κατά μέσο όρο 32.000 άτομα εκτοπίζονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Πάνω από 8.000 παιδιά πεθαίνουν από υποσυτισμό και περίπου 3.000 πεθαίνουν τη μέρα που γεννώνται. Έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τώρα, όχι αργότερα. Σήμερα, όχι αύριο. Γνωρίζω τι σημαίνει να ζει κανείς κατάσταση σειράξεως. Να μην έχει καταφύγιο. Να μην έχει τα βασικότερα. Να λύσει φόβο. Να ζει σε φόβο, συγγνώμη. Και να του έχει αφαιρεθεί η αξιοπρέπειά του. Ως παιδί και κατόπιν ως φοιτητής έζησα τα δεινά του λαού της Κύπρου. Των Ελληνοκυπρίων και των Τούρκοκυπρίων. Έζησα το πόνο της εξορίας. Κατάλαβα στο πετσί μου τη σημασία και την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να είμαι σαφής. Οι επιπτώσεις των σειράξεων δεν σέβονται εθνότητα ή θρησκεία. Φύγουν τους πάντες. Γέρους, νέους, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται σε ανάγκες, όχι πολιτικές σκοπιμότητες. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρομερές προκλήσεις στο εγγύς μέλλον. Πρώτα απ' όλα, θέλω να αποτίσω φοροτιμής ε, στους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και στην παροχή ανακούφισης. Κάθε μέρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλο, ανεξάρτητα από ταυτότητα, θρησκεία, εθνικότητα και ας φέρουμε στο μυαλό μας τη δολοφονία του Βρετανού εργαζόμενου στον ανθρωπιστικό τομέα David Haynes από το Ισλαμικό κράτος. Επίσης ας θυμηθούμε τη δολοφονία των, εκτά, των οκτώ θαραλέων ε, εργαζόμενων στην ανθρωπιστική, στην ανθρωπιστική βοήθεια και την υγεία που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τους κινδύνους του έμπολα. Αυτές είναι οι ε, οδυνηρές υπομνήσεις των κινδύνων που αντιμετωπίζουν αυτοί που εργάζονται για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά επίσης μας υπενθυμίζουν ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η παραβίαση των πιο βασικών θεμελιωδών αρχών που έχει καθορίσει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ο αριθμός των επιθέσεων κατά των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα έχει τετραπλασιαστεί από το 2003. Ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ευαίσθητος λόγω της αυξανόμενης ε, συχνότητας και εντάσεως των θεομηνιών σε αναπτυγμένε χώρες, ακόμη και στην Ευρώπη. Συμβαίνουν επίση, για παράδειγμα, οι πλημμύρες που είδαμε στα Βαλκάνια τον περασμένο Μάιο ήταν οι χειρότερε για 100 χρόνια στην περιοχή. Η συλλογική ανταπόκριση της Ένωσης σε αυτήν τη θεομηνία ήταν άμεση και εντυπωσιακή. 23 κράτη-μέλη έδρασαν αλληλέγγυα υπό το συντονισμό του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποστέλλοντας εμπειρογνώμονες και ζωτική σημασία βοήθεια. Πέρα από τις ε, ανθρώπινες τραγωδίες, οι θεομηνίες έχουν επίσης επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την ε, αύξηση. Η διαχείριση των κρίσεων σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τον όλο κύκλο των θεομηνιών, περιλαμβάνοντας την πρόκληση και την ετοιμότητα. Την πρόληψη, συγγνώμη, και την ετοιμότητα. Και το κάνουμε αυτό στα κράτη-μέλη μα, βοηθώντα τα να μειώσουν του κινδύνου, αλλά και διεθνώ στα πλαίσια του πλαισίου χιόγκο για δράση. Η επικείμενη παγκόσμια διάσκεψη τον επόμενο Μάιο στο Σεντάι θα είναι μια ευκαιρία η πρόληψη και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των θεμενιών να είναι ισότιμες προτεραιότητες με την ανταπόκριση στις θεομηνίες. Οι απόψεις του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές και είμαι διατεθειμένος να συζητήσω μαζί σας εν ώψη αυτής της συνδιάσκεψης. Στον τομέα των σειράξεων η κατάσταση είναι δραματική. Για πρώτη φορά έχουμε τέσσερις κρίσεις επίπεδου τρία που είναι η υψηλότερη ταξινόμηση στο σύστημα των ΗΠΑ Συρία, Ιράκ, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και Νότιο Σουδάν. Αλλά υπάρχουν και άλλες παρατεταμένες κρίσεις που εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, Παλαιστίνη, Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, Μαλή, Κολομβία, Μιανμάρ, για να αναφέρω μόνο κάποιε. Στη Συρία παρατηρούμε μία από τις μεγαλύτερε ε, ανθρωπιστικές καταστροφέ που έχουν σημειωθεί ποτέ. Πολύ πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν θυγεί από τη σύραξη. 6,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά είναι παιδιά, είναι εσωτερικά εκτοπιστέντες. Και ο αριθμός των προσφύγων έχει υπερβεί τα 3 εκατομμύρια. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα, όχι αύριο. Επιπλέον, έχουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της επιδημίας έμπολα στη Δυτική Αφρική. Η έμπολα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τεράστιας κλίμακας θεομηνία. Είναι σαν να είναι ένας τυφώνας σε αργή κίνηση και επίσης είναι απειλή στην ε, πλανητική ασφάλεια όπως την καθορίζει το Συμβούλιο Ασφαλή των Εθνών πίσω από τις ε, ανισχυτικές στατιστικές για την τρομερή επέκταση του ιού βρίσκονται πραγματικές ανθρώπινες ζωές, λαοί και κοινότητες που θα χρειαστούν και ψυχολογική βοήθεια μετά την ανάκαμψη. Αυτές είναι πιεστικές κρίσεις, παρούσες και χρειάζονται αμέσως απάντηση, αλλά επίσης και μακροχρόνιο σχεδιασμό αυτή η μοναδική κατάσταση έχει θέσει το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα υποτρομερή πίεση. Είμαι πεπισμένος ότι η παγκόσμια ανθρωπιστική συνάντηση κορυφής το 2016 θα συμβάλλει στην βελτίωση των δυνατοτήτων του διεθνού συστήματος να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη βοήθεια, βοήθειας. Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση δυστυχώς δεν συμβάλλει στην ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για τη σταθερή και αποφασισμένη δέσμευση για την υποστήριξη ουσιαστικών επιχειρήσεων που σώζουν ζωές. Είναι επιτακτικό να αποφύγουμε διακοπές στις δραστηριότητες οικονομικής βοήθειας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε... Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία επαρκή ροή πληρωμών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Και τέλος, ορισμένα λόγια για το όραμά μου. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, αλλά εξίσου μεγάλη είναι η αποφασιστικότητα και ο ενθουσιασμός μου. Θέλω να ολοκληρώσω την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Καταρχήν, θα συνεχίσουμε με, το κύριο, με την κύρια εντολή μας έτσι ώστε να χορηγήσουμε βοήθεια στα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να φτάσει με πολύ λίγα και πολύ αργά. Ούτε μία φορά θέλω να συνεισφέρω έτσι ώστε οι υπεύθυνοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να μπορέσουν να παραμείνουν και να παραδώσουν και δεν μιλώ μόνο για τις μεγάλες κρίσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά και για τις ξεχασμένες κρίσεις, όπως ονομάζονται. Δεύτερον, θα ήθελα να είμαι ο εκπρόσωπος των πλέον ευάλωτων, η φωνή εκείνων που δεν διαθέτουν φωνή. Θα εργαστώ την ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη, έτσι ώστε η φωνή εκείνων που πλήττονται να φτάσει στις τράπεζες λήψης αποφάσεων. Με θορύβησαν οι μαρτυρίες σε μια πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης για τη βία και την παρενόχληση των γυναικών της Συρίας που έχουν εκτοπιστεί. Οι γυναίκες και τα παιδιά βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και θα ήθελα να τους προσδώσω τη δέουσα προσοχή. Τρίτον, θα υπερασπιστώ τις ιδιαιτερότητες και τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει μία συλλογική βάση στην Ευρώπη, η συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σίγουρα η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανθεκτικότητα. Η επένδυση στην ε, ανθεκτικότητα είναι πολύ πιο σημαντική για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κρίση. Γι' αυτό θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Μίμικα, που είναι υπεύθυνος για θέματα ανάπτυξης. Πέμπτον, χρειαζόμαστε μία κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση έμπολα. Εργαζόμαστε στην Επιτροπή επί του θέματος μέσω του Κέντρου Συντονισμού Επίγουσας Ανταπόκρισης, ERCC, που συνδέεται με τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς εταίρους μέσα στα πλαίσια των μεγάλων χορηγών ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειλικρινά όμως τα αποτελέσματα δεν έχουν φτάσει. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Έκτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε προστατεύοντας τους Ευρωπαίους πολίτες. Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας πολιτικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πλέον αξιόπιστη και προβλέψιμη καθώς και αποτελεσματική απάντηση στις μεγάλες καταστροφές. Τέλος, σε σχέση με την συνεκτική προσέγγιση, θα συνεχίσω το έργο της προκατόχου μου. Είμαστε εντός αλλά εκτός. Γι' αυτό, εάν διοριστώ, θα συνεργαστώ με την ύπατη εκπρόσωπο και άλλους επιτρόπους για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη ρίζα της κακοδαιμονίας, και να μπορέσουν οι χώρες να επανέλθουν στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα συνεχίσω να διασφαλίζω την, τις πραγματικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να έχουν πρόσβαση στα θύματα και να μπορέσουν να τα βοηθήσουν. Τους το χρωστάμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρέθηκα σε βαθιά νερά εκπαίδευσης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, περιέχει πολλά θέματα επίγουσας ε, βοήθειας και αντιμετώπισης καταστάσεων κατεπήγοντος. Εάν ε, όμως επειδή μαθαίνω πολύ γρήγορα, σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι νύχθη για, για να κατανοήσω καλύτερα τα θέματα αυτά. Και θα έρχομαι πολύ συχνά στην Επιτροπή σας για να συζητώ αυτά τα ζητήματα μαζί σας. Ευχαριστώ. Um, thank you, Mr.